Az elnök Jó reggelt kívánok, kollégák! A mai... Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Έρχεται η συνεδρίαση. Ξεκινάμε με την πρώτη ψηφοφορία. Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Λόραντ Βίντσε ο οποίος ήθελε να μιλήσει ε, με βάση το άρθρο 59.4 για την αναπομπή στην Επιτροπή για τα προσωρινά μέτρα που αφορούν τα χρονικά όρια για την συλλογή και εξέταση σε σχέση με την επιδημία του κορονοϊού. Έχετε τον λόγο κύριε συνάδελφε. Καλημέρα σας. Έχουμε λοιπόν είχαμε την ψηφοφορία η οποία αφορούσε τα όρια του κανονισμού 788 της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών σε σχέση με το ξέσπασμα του κορονοϊού η οποία αποφάσισε να αναπεμφθεί το θέμα στην Επιτροπή ΑΦΚΟ σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 4. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. το αίτημα των, ε, του βουλευτή θα τεθεί σε ψηφοφορία μετά τα υπόλοιπα ζητήματα της ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία θα είναι από τις 9 μέχρι τις 10 και 4. Θα ακολουθήσουμε την ίδια μέθοδο όπως ε, και σε προηγούμενες ημέρες. Όλες οι ψηφοφορίες θα είναι ονομαστικές και τα αποτελέσματα αυτά θα δημοσιευτούν στην σελίδα της Ολομέλειας. Οι επεξηγήσεις ε, ψήφου μπορούν να υποβληθούν γραπτός, ε, κατ' εξαίρεση μόνο αυτές οι οποίες ε, περιέχουν 400 λέξεις maximum θα γίνουν δεκτές. Άρχεται η πρώτη ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε μέχρι τις 10 και 4 τα αποτελέσματα της ε, ψηφοφορία θα ανακοινωθούν 1 και 30. Σας ευχαριστώ. Az első napirendi pont megvitatására 9 óra 10. Το πρώτο σημείο τη ημερήσια διάταξη θα ξεκινήσει στι 9 και 4. Οπότε διακόπτουμε μέχρι τι 9 και 4. Καλημέρα. Ξεκινάμε. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι δήλωση της Επιτροπής που αφορά την αρπαγή γεών και αποψήλωση δασών στον Αμαζόνιο. Να ενημερώσω τα μέλη ότι για αυτή τη συζήτηση δεν υπάρχει διαδικασία catch the eye και δεν θα δεχτούμε μπλε κάρτες. Ευχαριστώ. Καταρχάς, να δώσω το λόγο στον κύριο Σίνκεβιτς, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Αμαζόνιος είναι ένα δάσος ε, που έχει μοναδική θέση, έχει μοναδικό ρόλο όσον αφορά την υγεία του πλανήτη μας, για τη βιοπικιλότητα και για το κλίμα. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το δάσος του Αμαζονίου για τους ηθαγενείς που είναι το σπίτι τους και εξαρτώνται από το δάσος για τη διαβίωσή τους και για τη συντήρηση του πολιτισμού τους. Οι προκλήσεις που επηρεάζουν την περιοχή του Αμαζονίου είναι περίπλοκες, πολυσχηδείς και χρειάζεται περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των χωρών που είναι, έχουν κοινή ιδιοκτησία τον Αμαζόνιο ε, ε, και είναι και κάτι που σχετίζεται και με κοινωνικο πτυχές και θέματα όπως η φτώχεια, η διαφθορά, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η κατάχρηση, η αστάθεια και η ασφάλεια. Οι περιοχές των αυτοχθόνων και των τοπικών κοινοτήτων στον Αμαζόνιο έχουν σύνορα με τα βασικά οικοσυστήματα της περιοχής. Οι τοπικές κοινότητες θα πρέπει να ανήκουν στη λύση. Η αντιμετώπιση της αποδάσωσης στον Αμαζόνιο είναι πολύ σημαντική, όχι για να καταπολεμηθεί το πρόβλημα όσον αφορά την ποικιλότητα στον κόσμο και αλλαγή του κλίματος, να πετύχουμε και βιώσιμη ανάπτυξη και την εκρίζωση της φτώχειας. Σύμφωνα με τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Πράσινη Συμφωνίας και τη νέα στρατηγική για το 2030 για τη βιοπικιλότητα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει το θέμα τη αποψήλωση των δασών και θέλουμε να ηγηθούμε όσον αφορά τη διεθνή προσπάθεια. Χρησιμοποιήσουμε εμπορική, πολιτική, διπλωματική ε, πολιτική και τα μέσα για την οικονομική ανάπτυξη. Σε παγκόσμιο επίπεδο θέλουμε να έχουμε φιλόδοξο παγκόσμιο στόχο με το 2020, σχετικό πλαίσιο και έχουμε το 2050 όλα τα οικοσυστήματα του κόσμου και τα δάση να αποκατασταθούν, να γίνουν ανθεκτικά και να προστατεύονται επαρκώ. Το παγκόσμιο πλαίσιο πρέπει να συμπεριμένει συγκεκριμένου στόχου για να μην χάνονται τα δάση και να διαφυλάσσονται τα οικοσυστήματα και η υγεία του, σύμφωνα με τι προτάσει στη στρατηγική βιοπικιλότητα τη Ευρωπαϊκή Ενώση. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε δράση κατά τη αποψήφιση των δασών και τη επιδείνου καταστάσεων των δασών, σε ένα μέρο εφαρμογή τη Συμφωνία των Παρισίων, συμπεριλαμβανομένη και συνεχή προσπάθεια να αυξήσουμε του φιλόδοξου στόχου για τα δάση σε εθνικό επίπεδο και να υποστηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών στα πλαίσια τη προσπάθεια μειώσεω τη ε, αποψήλωση των δασών και τη επιδείνωση τη υγεία των δασών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την αποψήλωση των δασών στα πλαίσια τη ανακοίνωση που κάναμε για να αυξήσουμε τι δράσει τη Ευρωπαϊκή Ενώση για να αποκαταστήσουμε τα δάση του κόσμου είναι μια απόφαση που υθετήσαμε τον Ιούλιο του 2019. Σαν πλαίσιο τη συνέχεια που δώσαμε στην ανακοίνωση την περσινή, θα παρουσιάσουμε το 2021 νομοθετικού περιεχομένου πρόταση και άλλα μέτρα, ώστε να αποφύγουμε ή να την, τη διάθεση προϊόντων που σχετίζουν την αποψήλωση των δασών, να μην διατίθεται στην αγορά τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και να προωθούμε εισαγωγέ φιλικέ ω τα δάση και κάνουμε αξιολόγηση συνεπειών σε αυτή τη φάση. Μέσα που συμπεριλαμβάνουν εθελοντικέ περιβαλλοντικέ δεσμεύσει τη βιομηχανία, υποχρεωτική ετικετοθεσία, η σωστή αντιμετώπιση, συστήματα πιστοποίηση, προσεγγίση σύμφωνα με το σύστημα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω που απαγορεύει και την παράνομη αλία, κάτι παρόμοιο, διμερή συμφωνία ή άλλα μέτρα. Καλωσορίζουμε τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για προσπάθειες καταπολέμησης οψίλωση των δασών και το σχέδιο νομοθεσία Burkhardt και τη σχετική έκθεση που αν υιοθετηθεί θα αξιολογηθεί προσεκτικά για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα τη αποψήλωση των δασών. Επίσης πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο να συνεργαστούμε το ιδιωτικό τομέα, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να έχουμε μεγαλύτερης προσπάθειας από πλευρά του ιδιωτικού τομέα για τα μέτρα αυτά. Όπω ανακοινώθηκε στη Στατική Βιοπικιλότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση θα υποβάλει μια νέα πρωτοβουλία το 2021 όσον αφορά τη βιώσιμη διακυβέρνηση των επιχειρήσεων. Θα είναι θέματα περιβαλλοντικά, ανθρώπινα δικαιώματα, ε, σωστή αντιμετώπιση ε, στου διάφορου τομεί. Άλλε δράσει. θέλουμε να δημιουργήσουμε πολυσχηδού πλατφόρμα για την αποδάσωση για την αουσία των δασών και θα συνεδριάσει αυτό ο φορέα τον Οκτώβριο και θα έχουν παρατηρητήριο που θα χρησιμοποιεί σχετικά δεδομένα για να διευκολύνει ανταλλαγή πληροφοριών για την αποψήφιση δασών στον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασισμένη να συνεργαστεί και να υποστηρίξει προσπάθειε ε, χωρών εταίρων στον Αμαζόνιο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ανθρώπινα δικαιώματα, κυρίω των αυτοχθόνων πληθυσμών και τοπικών κοινοτήτων στον Αμαζόνιο προστατευτούν και θέλουν προστατεύσουμε και το περιβάλλον. Αυτά είναι στο επίκεντρο των αξιών που ε, υποστηρίζουν τις σχέσεις με τρίτες χώρες, όπως είναι και οι χώρες της περιοχής του Αμαζονίου. Αυτά τα θέματα λοιπόν συστηματικά συζητούνται στο μηχανισμό του διαλόγου του πολιτικού συνεργασία. Ο διάλογος δεν περιορίζεται σε κεντρικές κυβερνήσεις. Επίσης, ενεργά συζητούμε με ευρύ φάσμα εμπλεκομένων φορέων. Σε υποεθνικό, σε τοπικό επίπεδο επίσης, με δικαστικές αρχές, κοινωνία των πολιτών, και με διάφορες ενώσεις επιχειρήσεων συζητούμε. Ο διάλογος αυτός είναι το κλειδί της επιτυχίας. Συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου με χώρες στην περιοχή είναι ένας άλλος τρόπος ούτως ώστε να προωθήσουμε τη συνεργασία σε διεθνείς υποχρεώσεις και προσπάθειες για το κλίμα και το περιβάλλον πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης. Τα κεφάλαια αυτά τα σχετικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με τα αίτια της αποξύσεως των δασών μέσω της βοήθειας της αναπτυξιακής Στηρίζουμε τα δάση, χρήση των γεών, βιώσιμη διαβίωση των διαφόρων πληθυσμών και έχουμε διάφορα προγράμματα που ανέρχονται τα προγράμματα σε 166 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Η προστασία τη βιοπικιλότητα, η καταπολέμηση οξύδου των δασών απαιτεί προστατευμένε περιοχέ και σωστή διακυβέρνηση. Επίση, συνάδει με τη βελτίωση τη διαβίωση των οπικών πληθυσμών και το σεβασμό των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση για βιώσιμη ανάπτυξη είναι στο επίκεντρο τη αναπτυξιακή μα στρατηγική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την εφαρμογή τη ε, της απόφασης 169 για του αυτόχους πληθυσμού του Διεθνούς Γραφείου Εργασία και την εφαρμογή των προσανατολισμών του ΟΗΕ για την κυβέρνηση ε, των αγορών ε, γεών και δασών και τη χρήση αυτών και έχουν χρησιμοποιήσει διάφορα μέσα για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων και για τους προασπιστές του περιβάλλοντος. Δυστυχώς, συχνάκης, ε, διακυβεύονται όλα αυτά στην περιοχή του Αμαζονίου. Προσβλέπω στενή συνεργασία μαζί σα Είναι σημαντικό το θέμα και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Πρώτος ομιλητής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είναι η κυρία Μακίνες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο που εξέφρασε την προσήλωσή του και τη δέσμευσή του για το μέλλον. Βέβαια αυτή τη συζήτηση την είχαμε και πέρυσι όταν βλέπαμε να καίγεται ο Αμαζόνης στο Κοινοβούλιο και δυστυχώ παρά τι ανησυχίε που εκφράσαμε δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εξού και ξανά είμαστε εδώ σήμερα για να συζητήσουμε την αρπαγή και την αποψήλωση των δασών. Δεν μπορούμε να πάψουμε να προσέχουμε το τι συμβαίνει εκεί. Υπάρχουν λοιπόν ε, τα προβλήματα της, ε, των εξαρκτικών δραστηριοτήτων ε, και της αρπαγής γεών που φαίνεται να νομιμοποιείται από την βραζιλιανική κυβέρνηση και έτσι ιδιωτικά χέρια θα πάρουν τις δημόσιες γέες, τα μεταλλεία και οι πυρκαγιές και όλα αυτά. Μιλάμε για 60 εκατομμύρια εκτάρια. Εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο επεξεργαζόμαστε νέες κλιματικές διατάξεις για να έχουμε το και ουδετερότητα μέχρι το 2050. Θέλουμε να είμαστε πρωτεργάτε, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και μόνοι μας. Είδαμε τις ε, αυξήσει, ε, μάλλον τις εκπομπές ε, στην Ευρώπη, τις εκπομπές του Ξύλου άνθρακα να μειώνονται στην Ευρώπη και λόγω της COVID, ενώ αυξάνονται στη Βραζιλία και λόγω της αποψήλωση. Επομένως, εξακολουθούμε να ανησυχούμε. Και σε ό,τι αφορά το άνοιγμα των αγορών μα, στο βόλιο κρέα ή στη σόγια από τη χώρα αυτή. Υποτίθεται ότι θα ενισχύσουν όλες αυτές οι διατάξεις και συμφωνίες ε, τη δέσμευση της χώρας υπέρ πιο περιβαλλοντικών μέτρων, όμως εμείς είμαστε επιφυλακτικοί, διότι έχουμε και τη δική μας ε, παραγωγή κρέατος ε, και θέλουμε πρωτεΐνες για να ταΐσουμε τα ζώα. Από πού έρχονται αυτές, έρχονται από τη Βραζιλία. Εμείς έχουμε επιβάλει κανόνες στα δικά μας τα, τα κράτη, αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται με τα εισαγόμενα προϊόντα. Θέλουμε επίσης ε, να προωθήσουμε την ε, νομοθεσία περί βιοπικιλότητα και έχουμε και την εμπορική νομοθεσία, τι πρωτοβουλίε που μόλις δρομολογήθηκαν. Βλέπουμε να υπάρχει μεγάλη αντίφαση ε, μεταξύ πολιτικών, γεωργικών, εμπορικών πολιτικών. Πρέπει όλα αυτά να ευθυγραμμιστούν, να αρμονιστούν το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ, η πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βαν Μπρέντ, εκ των Σοσιαλιστών είναι η επόμενη. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο. Ε, μου άρεσε η εισαγωγική σας παρέμβαση. Εγώ δεν αμφιβάλλω για τις προθέσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει ε, το πρόβλημα του κλίματος σε συνδυασμό με την αποψήλωση. Αλλά αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας, που ξέρετε ποιοι είναι, είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό, είναι κομβικό να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στον Αμαζόνιο, που είναι μεγαλύτερη δεξαμενή άνθρακα στον πλανήτη και το δραματικό είναι ότι αλλάζει. Αλλάζει η κατάσταση και μόνο αν δράσουμε αποφασιστικά μέχρι το 2030, ε, ουσιαστικά θα έχει αντιστραφεί κατάσταση και θα είναι καθαρός εκπομπός διοξιδίου του άνθρακα ο Αμαζόνης. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να δράσουμε τώρα. Ε, σίγουρα ε, δεν είναι ακόμη τα πράγματα ε, τόσο καταστροφικά ώστε να μην μπορούμε να έχουμε ε, κάποια τύχη. Πάντως κάθε μήνα τα πράγματα επιδεινώνονται. Ακόμα δεν έχει καν ξεκινήσει η εποχή των πυρκαγιών. 80% της υποψήλωσης συνδέεται με τη γεωργία και με την κατανάλωση στην Ευρώπη. Άρα και εμείς έχουμε να κάνουμε ε, δουλειά εδώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ένα στόχο. Πρέπει να επαγρυπνούμε. Η κυβέρνηση Μπολσονάρο χρησιμοποιεί την κρίση της COVID-19 για να πιέσει προς περισσότερη απορρίθμιση στην περιβαλλοντική νομοθεσία. Και ήδη γνωρίζουμε ότι ε, το 30% ε, του προϋπολογισμού της Εθνικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος ε, θα διατεθεί για πυροσβεστικές δράσεις. Και υπάρχει το θέμα της παράνομης υλοτομίας ε, ο επικεφαλής επιστητής διαστημικής υπηρεσίας ε, ε, συλλέγει κάποια στοιχεία για την αρπαγή γεών και συλλέγει κάποια στοιχεία τώρα μέσω των και για την υποτίθεται για να δει τι γίνεται με την, σε επιπτώσεις της COVID-19. Είπατε ότι πρέπει να έχουμε ε, μια ασφαλιστική δικλίδα σε συμφωνίες, ε, την περιβαλλοντική δηλαδή ρήτρα για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Στην περίπτωση της Βραζιλίας έχουμε υπογράψει ένα χρόνο. Η κατάσταση επιδεινώνεται. Μπορούμε να την πιστέψουμε τη Βραζιλία επομένω. Άρα το Κοινοβούλιο πρέπει να ζητήσει πραγματικέ διασφαλίσει σε ό,τι αφορά τον Αμαζόνιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα καθορίσει και τι συζητήσει για την εμπορική συμφωνία. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα σα τα πω ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν μπορούμε να δεχθούμε ελεύθερο εμπόριο χωρί κλιματική δράση. Και αν θέλουν οι άλλες χώρες να είναι εμπορικοί μας εταίροι, πρέπει να είναι εταίροι μας και στην περιβαλλοντική δράση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις συζητήσεις που θα έχουμε στο μέλλον και για την μελλοντική πολιτική. Και το λέω ξεκάθαρα αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Κάνιας από την ομάδα Renew. Ευχαριστώ πολύ. Ο Αμαζόνιος ε, κινδυνεύει. Έχουμε αρπαγή γεών, υλοτομία και εμπρισμούς ε, για γεωργικές ε, δραστηριότητες και μεταλλεία εξοριστικές δραστηριότητες. Αυτό έχει να κάνει με, έχει ως αποτέλεσμα τεράστιες εκτάσεις να αποψηλώνονται. Ποια είναι η στρατηγική για να ανατραπεί αυτή η πολιτική που απειλεί το κλίμα, τη βιοπικιλότητα αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη των χωρών του Αμαζονίου και απειλεί και τα δικαιώματα των πολιτών των χωρών να έχουν αξιοπρεπή ζωή ο νεοπικιακρατικός πατερναλισμός είναι σωστός ή θα έπρεπε ίσως να έχουμε μια σωστή στρατηγική με σεβασμό, με δεσμεύσεις συνεργασία και ε, συμφωνίες ουσιαστικά. Γιατί αν θέλουμε να έχει παγκόσμιο και πραγματικό αντίκτυπο η δική μας στρατηγική. Χρειαζόμαστε εταίρους που θα ακολουθήσουν τη στρατηγική μας... και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο με βάση δεσμευτικών ε, συμφωνιών. Αυτό ζητούμε και υπαγρυπνούμε ως Κοινοβούλιο Βλέπουμε ότι κάποιες χώρες με αποφάσεις πηγαίνουν στη λάθος κατεύθυνση, όμως υπάρχουν και θετικές ε, διατάξεις. Έχουμε χώρες που έχουν υπογράψει ε, τη Συμφωνία των Παρισίων και άλλες περιβαλλοντικές συμφωνίες. Ε, οπότε μπορούμε, πιστεύω, να βοηθήσουμε χώρες οι οποίες πλήττονται και έχουν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες οικονομικές και κοινωνικές. Πρέπει να προστατεύσουμε τους αυτόχθονες, τους υπερασπιστές του περιβάλλοντος. Δεν είναι μόνες οι χώρες απέναντι στις κυβερνήσει τους. Ε, οι κυβερνήσεις όπως και εμείς αλλάζουν, ε, περνάνε ε, και η κατάσταση εκεί παραμένει, το περιβάλλον παραμένει και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και το πιο ισχυρό εργαλείο που έχουμε είναι εμπορικέ συμφωνίες και συμφωνίες σύνδεσης που είναι πολύ σημαντικές για τη συνεργασία με τους εταίρους μας, για την στρατηγική μας όπως είναι η συμφωνία της Ένωσης με τις χώρες Μερκοσούρ. Περιλαμβάνει κεφάλαιο για τη βιώσιμο περιβάλλον και είναι δεσμευτικό και το στοιχείο της στήρησης ε, της Συμφωνίας ε, του Παρισιού. Επομένω, δεν θα σβήσουμε τις πυρκαγιές, ούτε θα κλείσουμε τα μεταλλεία, ούτε θα σταματήσουμε την αποψήλωση με κηρύγματα και παρτερναλισμό, αλλά μόνο με συνεργασία και συμφωνίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα δίνω τον λόγο στην κυρία Πένιε, εξ ονόματος της ομάδας ID. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ρεκόρ ε, η αποψήλωση και παγκόσμιο, παγκόσμια συγκίνηση και το δέος ε, που προκαλείται ε, και στα τροπικά δάση και στα κανονικά. Εσείς συζητάτε εδώ πέρα, αλλά βλέπουμε να υποβαθμίζονται οι αγροτικές γιές, αλλά όχι μόνο στην Βραζιλία, αλλά και εδώ. Ποιος στέει ε, στη Γαλλία βλέπουμε πολύ μεγάλο τέτοια ποσοστά. Ε, φταίει το μοντέλο το γεωργικό ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς στρέφετε τα βλέμματα στην Βραζίλικα, και στο Αμαζόνιο, αλλά έχετε ευθύνες εδώ. Υπάρχουν πρακτικές τρίτων χωρών, αλλά η αποψήλωση ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο εμεί προκαλούμε, γιατί παίρνουμε ξύλο, εισάγουμε παράνομο ξύλο τι γίνεται με το φίνικελο, το κακάο, το καουτσούκα και τη σόγια. Σε ό,τι δεν αφορά τι αρπαγέ γεών, είναι σαφέ το πρόβλημα. Πρόκειται για τη γεωργική παγκοσμιοποίηση. Γιατί η σόγια, η καλλιέργεια τη σόγια στην Αμαζόνια είναι το βασικό ε, αίτιο τη ε, αποψήλωση. 70-80% τη σόγια ουσιαστικά χρησιμοποιείται για να θρέψει ε, ζώα ε, τη κτηνοτροφία. Και ε, αυτό το μοντέλο, το εντατικό μοντέλο ε, είναι δική μας ε, ευθύνη. Έχουμε επίσης αυτές τις συμφωνίες. Η τελευταία επονίδη συμφωνία είναι αυτή με τις χώρες Μερκοσούρ. Όταν ενθαρρύνονται τέτοιες πρακτικές με τις χώρες Μερκοσούρ είναι ντροπή, πώς θέλουμε να συνετίσουμε τη Βραζιλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει από την Νότια Αμερική πάνω από 300.000 ε, τόνους ε, να εισαγάγει με μειωμένους ε, δασμούς. Έχετε αυτή τη φιλοευρωπαϊκή πολιτική που ουσιαστικά σας οδηγεί να είστε μοιραία και ένας κρίκος αυτής της καταστροφικής αλυσίδας πολλοί από εσά δουλοπρεπώ ε, υπογράφετε όλε αυτέ τι εμπορικέ συμφωνίε που ουσιαστικά οδηγούν σε μεγαλύτερη αποψήλωση. Πρέπει να βγούμε εκτό αυτών των συμφωνιών ε, που έχουμε επικυρώσει, να πάψουμε να εισάγουμε αυτά τα προϊόντα και να παίρνουμε προϊόντα από τα γεωργικά αγροκτήματα ε, τη περιοχή μα. Να προχωρήσουμε σε ένα μοντέλο ηθικό. Ευχαριστώ τον λόγο, κυρία Καβατσίνη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου με του ανθρώπου στον Αμαζόνιο και ειδικά στη Βραζιλία που υποφέρουν ε, από τον COVID-19 και χάνουν του οικείου του. Τι μπορεί να είναι πιο σοκαριστικό στην κατάσταση αυτή από το να ακούμε έναν υπουργό να λέει ότι δεν χρειαζόμαστε περιβαλλοντική προστασία τη στιγμή που όλοι ασχολούνται με τον κορονοϊό. Αυτό τον έπιασα να λέει στο βίντεο τον Βραζιλιανό Υπουργό. Η αποδάσωση αυξάνεται και αυτό είναι άμεση συνέπεια συνέπειών της κυβέρνησης. Ε, διαλύουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, σταματάν τα πρόστιμα για την λαθροϊλοτομία και επιπλέον η κυβέρνηση Μπολσονάρου υποστηρίζει ένα νόμο περί αρπαγής γης που μπορεί να ψηφιστεί ανα πάσα στιγμή. Εγώ θα στηρίξω οποιονδήποτε αντιμάχεται σε αυτά επί τόπου και ζητώ από του συναδέλφου μα στο Κογκρέσο τη Βραζιλία να μην ψηφίσουν τον νόμο περί αρπαγή. Αλλά και εμεί στην Ευρώπη έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε. Τα σούπερ μάρκετ στο Ηνωμένο Βασίλειο απειλούν να μποϊκοτάρουν τα αγροτικά προϊόντα τη Βραζιλία εάν περάσει ο νόμο. 350.000 άνθρωποι υπέγραψαν στην Γερμανία αυτή τη στιγμή μια αίτηση ζητώντας να γίνει το ίδιο. Πρέπει λοιπόν να σταματήσει από αποδάσωση και να σταματήσουμε να εξαρτώμαθε από το έδαφος. Και βεβαίως η Μερκοσούρ έχει πεθάνει. Είχε πριν μεγάλη αντίσταση αλλά πλέον ε, δεν βλέπω να υπάρχει κάποια πιθανότητα συμφωνίας με τη Μερκοσούρ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακολουθεί ο κύριος Τζαμπάσκη από το ECR. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, λοιπόν, αυτό το οποίο βλέπουμε Δυστυχώ ε, υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα και δεν ε,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 Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα ξεκινήσω από την αρχή. Για μία ακόμη φορά. Πάλι λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή έρχεται σε λάθος στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκλονίζεται ε, υπάρχουν άνθρωποι, εκατομμύρια που χάνουν ε, τις δουλειές τους, ε, ξαναγράφεται η ιστορία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται με τον Αμαζόνιο. Με τον Αμαζόνιο. Ο Αμαζόνιος δεν διέρχεται από καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι φόροι των ψηφοφόρων σας δεν πηγαίνουν στον Αμαζόνιο. Η συζήτηση αυτή είναι άχρηστη. Δηλαδή, Ας συζητήσουμε και αν υπάρχει νερό στον Άρη. να μπει στην ημερήσια διάταξη. Ζητάτε εδώ πέρα σαφήνια ιδεών και ταυτόχρονα τι γίνεται με τον αέρα. Μιλάτε για καθαρό αέρα και μετά έχουμε φορτηγά που διασχίζουν την Ευρώπη. Πρέπει να μιλήσουμε για τον καθαρό αέρα. Τώρα λοιπόν διδάσκουν οι άλλες ήπειροι το πώς καθαρίζει ο αέρας. Ή διατηρείται καθαρός. Αν ψηφίζει κανείς υπέρ της ρήπανσης του αέρα, ε, τότε δεν έχει δικαίωμα να μιλάει για τον Αμαζόνιο αλλά και στις ζούγκλες του Αμαζονίου ακούσαμε για την απεικιοκρατία, το προνόμιο των λευκών, να ζητήσουμε συγνώμη ότι υπάρχει ιστορική ευθύνη κτλ. Αγαπητοί συνάδελφοι, εάν θεωρείτε ότι θα πρέπει να αυτομαστιγώνεστε και ότι όλα αυτά θα σχεδίσουν ψήφους, κάνετε λάθος. Εάν θεωρείτε ότι δικαιολογώντας τις βάρβαρες αυτές πράξεις θα έχετε στήριξη, όχι δεν θα συμβεί αυτό. Όταν τελειώσει το πλιάτσικο θα έρθουν σε εσά. Και το δείχνει η ιστορία. Όλες οι επαναστάσεις έτσι ξεκινάνε. Αν θυμάστε το σφυροδρέπανο, ξεκινάνε από πλιάτσικο και μετά καταλήγουν μπολσεβίκοι. Δείτε και τι έγινε στη χώρα μου. Οπότε πρέπει να θυμόμαστε ότι τι νομίζετε, θα έχετε περισσότερες ψήφους. Όχι, όχι. Δεν θα υπάρχει άλλη βαρβαρότητα και διαγραφή της ιστορίας. Αν έχετε ε, ερωτήσεις ε, και ζητήματα για το απεικιοκρατικό παρελθόν, κάντε το. Αλλά μην ασχολείστε με εμά να ζητήσουμε εμεί συγγνώμη για κάτι για το οποίο δεν είμαστε ευθύνοι. Οι Βούλγαροι δεν γονατίζουν, οι Βούλγαροι ποτέ δεν ταπεινώθηκαν, οι Βούλγαροι δεν ζητάνε έλεος. Όταν μπαίνει κάποιος να κάνει πλιάτσικο, δεν του ανοίγουν την πόρτα. Στεκόμαστε όρθιοι και παλεύουμε και προστατεύουμε την πατρίδα μας, τον πολιτισμό μας, την οικογένειά μας. Έτσι κάνουμε. Σας εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία στην προστασία των δασών του Αμαζονίου. Πρόκειται για μια επική συζήτηση πλανητικών διαστάσεων και όταν θα έρθει η επόμενη παραδείγματος χάρη αν χρειάζεστε παραδείγματος χάρη ε, περισσότερους ε, περισσότερες ανεμογεννήτρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έρθω να το συζητήσουμε και υγεία εύχομαι Ευχαριστώ Απ' την ΚΟΕ τώρα η κυρία Χάζεκαμπ Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε Ο κόσμος είχε συγκλονιστεί πριν από λίγο καιρό από τις πυρκαγιές στον Αμαζόνιο και φαίνεται ότι όλα αυτά εκτοπίστηκαν από τις ειδήσει ε, από τον COVID, αλλά ε, δεν σταμάτησαν να συμβαίνουν. Έχει τεράστια σημασία ο Αμαζόνιος και για το κλίμα και για τον άνθρωπο και τα ζώα που κατοικούν εκεί. Οπότε ε, και με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Αμαζόνιος καταστρέφεται πάρα πολύ γρήγορα. Αυτά γίνονται για να γεμίσουμε τον τεπόζιτο των αυτοκινήτων και τα στομάχια μας. Και κάθε χρόνο εισάγει η Ευρώπη 1,5 εκατομμύριο τόνους σόγια και ε, 400.000 τόνους βοδινού κρέατος. Εάν λοιπόν θέλουμε να σώσουμε τον Αμαζόνιο και θέλουμε να σταματήσουμε την απώλεια της βιοποικιλότητας πρέπει να κάνουμε κάτι. Κύριε Επιτροπέ, δεν θα έχετε στρατηγική με την βιοπικιλότητα όταν οι συνάδελφοί σας ταυτόχρονα ασκούν αυτήν την πολιτική γεωργίας και εξωτερικού εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν λέτε ναι κατά μιας πιστικής πολιτικής βιοπικιλότητας. Είστε διατεθειμένοι να πείτε ένα όχι, όχι στην καταστροφή του Αμαζονίου, στην εισαγωγή σόγιας για ζωοτροφή στην κατάργηση των επιδοτήσεων για την προώθηση του κρέατος. Να τρώμε λιγότερο κρέας. Αυτό δεν είναι καλύτερο μόνο για τον Αμαζόνιο, αλλά και για τα ζώα τα ίδια που τρώμε. Και ακριβώς αυτή τη στιγμή έχει την ευκαιρία να κάνει κάτι το Κοινοβούλιο. Απευθύνω έκκληση στους συναδέλφους να ξεκινήσει μία επιτροπή που θα διερευνήσει τα ζητήματα μεταφοράς των ζώων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Λεωνόρα Εύη από τους ΜΚΙ γραμμένους έχει τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Animal λικουαλίτη ΜΚΟ έδειξε τη διασύνδεση μεταξύ τη αποψίωση των ασθενών στην Αμαζονή και δημιουργία μεγάλων κτηνοτροφικών εκτάσεων που προορίζονται για ασφαγή και σχεδόν 6.000, 6.000 χιλιόμετρα ε, περίπου 60 ε, γήπεδα ε, την ώρα καταστρέφονται. Μια έκθεση τη Greenpeace για ότι σφαγιάζονται τα δάση, είναι ο τίτλο, λέει ότι οι καταναλώσει τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω συνδέονται με το 10% τη αποψήλωση των δασών στον κόσμο. Οι Ευρωπαίοι πολίτε ε, είναι και αυτοί συνένοχοι και έχουν επίγνωση τη καταστροφή ε, των πολιτήμων εικονισυστημάτων στον πλανήτη, όπω είναι η Αμαζόνιο. Και λυπάμαι, από τη μία πλευρά έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει μια πρόταση νομοθετικού να περιεχομένου εγγυηθεί ότι τα προϊόντα που διανέμονται στι ευρωπαϊκέ αγορέ δεν θα συνδέονται με την αποψήλωση των δασών. Από την άλλη πλευρά, όμω, γίνονται διαπραγματεύσει όσον αφορά την εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκή Ενώσεω και Μερκοσούρ, αγνώντα την υποχρέωση τη νομική να εξασφαλίσετε ότι η συμφωνία δεν θα οδηγεί σε επιδείνωση κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μα πει με ποιο τρόπο προτίθεται συγκεκριμένα να αντικατοπτήσει τι δεσμεύσει που αναλήφθησαν για την προστασία των οικοσυστημάτων και την μείωση τη αποψή των δασών και στι εμπορικέ συμφωνίε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Άνλαμ Γιαρούμπα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Η αποψήλωση των δασών του Αμαζονίου συμβαίνει πολύ συχνά ή μάλλον συζητιέται πολύ συχνά. Το συζητήσαμε ήδη το θέμα το Σεπτέμβριο συζητήσαμε το πώς μπορούμε να σταματήσουμε τις πυρκαγιές που καίγουν ε, δάση που είναι οι πνεύμονες του κόσμου. Ταυτόχρονα προχωράμε προς εμπορική συμφωνία με τη Μερκοσούρ, χρησιμοποιούμε διπλωματικά μέτρα, ελπίζοντας ότι θα πιεστούν οι χώρες αυτές για να τηρήσουν τη Συμφωνία των, Παρισίων και να μειωθεί η απόψη των δασών. Επίτροπε, σωστά είπατε, ότι το σταμάτημα της αποψήρωσης των δασών είναι σημαντικότατο στοιχείο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή ε, Πολιτική Επικοινότητα και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Αλλά αν θέλουμε να είναι ανταγωνιστική η Ευρώπη και να παραμείνει ανταγωνιστική, πρέπει να επιβάλλει κάποιε απαιτήσει σε εμπορικού εταίρου. Στόχου του κλίματο, Φερρυπίν. Βιώσιμοι στόχοι θα πρέπει να ε, τίθενται. Οι εμπορικέ διαπραγματεύσει είναι ένα θέμα. Αλλά διάφορου αρμογή ε, όσον αφορά την εκπομπή άνθρακα θα ήταν ένα σημαντικό εργαλείο. Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι θα θυμόμαστε την ευημερία των ζώων, την ασφάλεια των τροφίμων, όλα αυτά τα πρότυπα και προδιαγραφές και αυτές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις συμφωνίες, διότι με αυτά τα πρότυπα αυτά είναι τα ίδια πρότυπα που δεσμεύουν του Πολωνού και του Γάλλου γεωργού. Ναι, για τι συμφωνίε, αλλά όχι στον αθέμητο ανταγωνισμό όσον αφορά τη γεωργία. Και όχι όσον αφορά του κινδύνου για την υγεία μα, όσον αφορά τα τρόφιμα παράγονται που δεν έχουν επιστοποιημένη ποιότητα. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος από τους σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Βαθιά στον Αμαζόνιο ζουν οι Τούνα, οι Τατά, οι φιλοί αυτοί αυτοχθόνων η περιοχή τους είναι θεωρητικά προστατευόμενη. Στην πράξη εισχωρούν εκεί πέρα κτηνοτρόφοι, υλοτόμοι και ορυχεία χρυσού. Ήδη υπάρχουν διάφοροι νόμοι που έχουν περάσει ή προγραμματίζονται από την κυβέρνηση Μπολσονάρου για να διευκολύνουν την εκμετάλλευση της γης ε, ή την αμνηστία στην κλοπή γης. Πρόκειται για μια κλοπή αλλά και οικολογική καταστροφή στον Αμαζόνιο όπου καταστρέφεται ο πνεύμονας με τον οποίο θα πολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Αλλά και η Ευρώπη έχει ευθύνη γιατί 10% της ε, καταστροφή των δασών οφείλεται σε εμά στην κατανάλωσή μας. Γιατί τρώμε σόγια, κρέας και καουτσούκ. Πολλές επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόβλημα και προσπαθούν να κάνουν μια παραγωγή πιο βιώσιμη. Πρέπει λοιπόν να βρούμε κάποιες απαντήσεις. υπέβαλα αυτή την εβδομάδα το σχέδιο έκθεσή μου σχετικά, το οποίο αφορά ακριβώ επιχειρήσει οι οποίε θέλουν να φέρουν κάποια προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι τράπεζε που του στηρίζουν θα πρέπει να δώσουν πολύ περισσότερη προσοχή στι συνθήκε παραγωγή. Χρειάζεται λοιπόν κάποια υποχρέωση, να υποχρεώσουμε τι εταιρείε να μην καταστρέφουν τα δάση, τα οικοσυστήματα ή να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και η κοινότητα των Ιτούνα Ιτατά θα ωφεληθεί από αυτή την κατάσταση. γιατί βεβαίως καταναλώνται προϊόντα στην Ευρώπη που καλλιεργούνται στη γη τους. Οι Ιτούνα οι Τατά δεν μπορούν να βασίζονται στην κυβέρνησή τους και στο ότι θα παρέμβει κατά της αρπαγής γης. Εξάλλου έχουμε ένα εξασθενημένο σύστημα δικαιοσύνης ή όπως στη Βραζιλία δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Θα πρέπει λοιπόν αν δεν το κάνουν οι ευρωπαϊκές εταιρείε να τις αναγκάσουμε με αστική ευθύνη, αλλιώς δεν γίνεται. Η τούρα, η τατά φαίνονται πολύ μακρινοί, αλλά η προστασία τους ε, εξαρτάται από τα προϊόντα που έχουμε στο σούπερ μάρκετ μας. Ας τα κάνουμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Νικόλα Στεφανούτα λοιπόν, κατόπιν από το Ρνιού. Μεταξύ των καλών και κακών ηγετών. Σε μια περίοδο κρίσεως πρέπει να κάνουμε διάκριση, πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες. Πρέπει να δούμε ποιες είναι, ποια είναι τα συμφέροντα του πληθυσμού ε, μακροπρόθεσμα ή μικρή ομάδα βραχυπρόθεσμα. Οι ηγέτες που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών πιστεύουν στη συνωμοτική θεωρία και παίρνουν αποφάσεις ε, με έναν τρόπο ενστικτόδη, όπως ο Μπολσονάρο ε, οι Βραζιλιάνοι φοβούνται για το αύριο, διότι χίλια άτομα πεθαίνουν την ημέρα από τον COVID-19 και ο Μπολσονάρο τι σκέφτεται τα συμφέροντα διαφόρων ομίλων επιχειρηματικών, κάποιων ομάδων επιχειρηματιών και δεν σκέφτεται καθόλου το συμφέρον του πλανήτη, ούτε το συμφέρον των Βραζιλιάνων πολιτών, ούτε του δάσους του Αμαζονίου. Το δάσος του Αμαζονίου θα αντιμετωπίσει καταστροφή η εποχή των πυρκαγιών ακόμα των δασικών δεν έχει ξεκινήσει. Θα δούμε τον πλανήτη να καίγεται σε λίγο. Η Βραζιλία κάνει βήματα οπισθοδρόμησης πολύ γρήγορα στον αφορά το περιβάλλον και προτάθηκε νέο νομοσχέδιο για να δίδονται τίτλοι ιδιοκτησίας σε γεωργούς που παράνομα κατέχουν γεές ε, αυτοχθόνων πληθυσμών. Τα στοιχεία δεν ψεύδονται. Πάνω από 90% Πέρσι ήταν παράνομε οι αρπαγέ γεών, οι αποκτήσει γεών ε, και κυρίω αφορούσε αρπαγέ γεών στην περιοχή του Αμαζονίου. Στα δύο λεπτά που έχω στη θέση μου, πρέπει στα 6 εκτάρια εξαφανίστηκαν στα δύο λεπτά που μιλάω εγώ στο δάσο του Αμαζονίου. Και 54 εκτάρια δάσου έχουν εξαφανιστεί σε όλο τον κόσμο σε αυτό το διάστημα. Συμφωνώ με την εισηγήτρια, την κυρία Μπόρκχαρτ, ότι θα πρέπει να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα και εδώ. Διότι και εμεί αποτελούμε τμήμα του προβλήματο. Δεν συμβαίνει μόνο στα δάση του Αμαζονίου. Υπάρχουν μικρά δάση τύπου Αμαζονίου και στην Ευρώπη θα πρέπει να επιληφθούμε του θέματος και θα πρέπει να βρούμε μια λύση τώρα ε, όταν δεν είναι ακόμα πάρα πολύ αργά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Κάμπο Μανώζη. Έχει, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους σας. Εγώ θα επιστρέψω στην πόλη μου σήμερα. Αύριο θα συναντήσω δημάρχους, επιχειρηματίες, εργαζομένους, βιοτέχνες. Κάποιοι θα με ρωτήσουν, Μάρκο, τι κουβεντιάσατε χτες στις Βρυξέλλες. Μιλήσατε για να, πώς θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις, πώς θα βγούμε από μια κρίση που θα είναι καταστροφική. Όχι. Θα απαντήσω ότι αφιερώσαμε όλο το πρωινό συζητώντας για τον Αμαζόνιο. Αλλά μιλήσατε για την αρπαγή υγειών, για την Κίνα. Όχι. Μιλήσαμε για τον Μπολσονάρο. Όχι. Αυτό το κοινοβούλιο αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο προφανώς επικεντρωνόμενο επί των επικρίσεων έναντι ηγετών συντηρητικών σε όλο τον κόσμο. Το είδαμε τι στάση είχαμε έναντι του Τραμπ και τι στάση έχει έναντι νομίμων κυβερνήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι η Πολωνία και η Ουγγαρία. Είδαμε σήμερα και διάφορες αναφορές στον Μπολσονάρου σαν τα προβλήματα στον Αμαζόνιο να ξεκινάνε και να γεννιόνται από αυτή την κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που μεταξύ άλλων είχε μεγάλα προβλήματα και δυσκολία όσον αφορά τη διαχείριση της ε, πανδημίας, όπως όλοι μας. Η νεοπικιακή στάση διαφαίνεται. Εμείς πώς το βλέπουμε, εμείς Ευρωπαίοι που κάνουμε, συνάπτουμε με το Βιετνάμ με εμπορικέ συμφωνίες που έχει περιβαλλοντικές προδιαγραφές πολύ πιο χαμηλές από αυτές των νοτιοαμερικανικών χωρών. Και το κόμμα μου, η ομάδα μου επικρίνει σοβαρά και την εμπορική συμφωνία με το Μερκοσούρ που ευτυχώς λόγω των Νοτιοαμερικάνων θα καταρρεύσει, δεν υπάρχει συνένεση και είναι ένα εμπορικό μοντέλο που αντιπροσωπεύει που έχει ξεπεραστεί αλλά δυστυχώς ο Επίτροπος Χόγκαν μας λέει ότι τώρα θα προχωρήσουμε θα προχωρήσουμε ίσια σαν να μην τρέχει τίποτα. Η υποκρισία λοιπόν από την πλευρά μας που είναι, είναι κρίμα εγώ πρέπει να παίξω το ρόλο του κακού. Πρέπει να παρουσιάζουμε θέσεις. Αυτή η στάση όμως είναι εις βάρος όλων. Και θα ζητήσουν να δώσουμε διαφορετική προσοχή οι πολίτες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον, ε, στην κυρία Μπρικμόν. Ευχαριστώ. Το 2020 αποψήλωση ρεκόρ στη Βραζιλία, καταπάτηση δικαιωμάτων των αυτοχθόνων, κίνδυνος για την ιδιοκτησία. Και είναι τόσο τραγική η κατάσταση στη Βραζιλία που αρχίζει να ξεσηκώνεται η Ευρώπη, θα υπάρξει μποϊκοκατάρισμα βραζιλιάνικων προϊόντων. Αλλά πρέπει να δούμε και τι έγινε και με τη Συμφωνία Μερκοσούρ. Η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ εμπόριο ε, ελαχιστοποιεί ε, ή προσπαθεί να υποτιμήσει τον αντίκτυπο όλων αυτών. Και εσείς, Επίτροπε, είπατε ότι ε, δεν είναι υπερβολική η κλιματική στόχη και μπορούν να επιτευχθούν. Αυτή η πράσινη διπλωματία, πού η πρασινη πλωματεια γιατί εγώ δεν τη βλέπω στην εμπορική πολιτική. Αν θέλουμε να εφαρμόσουμε τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, Συμβούλια και Κομισιόν πρέπει να καταγγείλουν και να ζητήσουν την ακύρωση του νομοσχεδίου στην Βραζιλία που στρέφεται εναντίον των δικαιωμάτων αυτοχθόνων και να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Να αναγνωρίσει επίσης ότι δεν πληρούνται οι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί στόχοι με τη Συμφωνία Μερκοσούρ. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Λούντγκρεν. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη παλαιότερα έβλεπε ότι κάθε λεπτό δύο γήπεδα ε, ισοδύναμη έκθαση στον Αμαζόνιο χανόταν. Έπειτα δημιουργήθηκε αυτό το σύστημα ε, για να μετράτε και να υπολογίζετε η απώλεια. Το 30% των δασών του Αμαζονίου Ουσιαστικά, μετά από, τους, ε, από τις πυρκαγιές ε, ήταν καλυμμένο από μία ε, και πάρα πολλά ζώα έχουν καεί με τις πυρκαγιές. Ουσιαστικά εξαφανίζεται σιγά σιγά το δάσος. 55% αύξηση της αποψήλωσης τους πρώτους μήνες ε, του 2020 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Καταστράφηκαν πάνω από 1.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δύο φορές η πόλη του Γκέτεμπορκ. Από τότε που να, μετρούν ε, τον Αύγουστο του 2015 έχουν καταστραφεί τεράστιες εκτάσεις και ο λόγος είναι ότι θέλουν να έχουν ε, οι αγρότες περισσότερες γιές για να καλλιεργήσουν ε, προϊόντα που χρησιμοποιούμε εδώ στην Ευρώπη, όπως το φινικέλαιο. Άρα εμείς συνεισφέρουμε στην αποψήλωση. Γιατί μιλάμε. Μιλάμε για περιβαλλοντικά περιβαλλοντικά καύσιμα. Άρα ακόμα πιο πολύ φινικέλαιο. Θέλουμε επίσης φιλοπεριβαλλοντικά καύσιμα και για τις αεροπορικές μεταφορές. Πάλι πιο πολύ φινικέλαιο θα απαιτήσει αυτό. Πραγματικά είναι αποφάσεις αυτές που δεν γίνονται αντιληπτές. Δεν γίνονται αντιληπτές από τον κόσμο. Έχουμε αυτές τις φιλοπεριβαλλοντικές δημόσιες συγκοινωνίες στην Σουηδία για τις οποίες καυχόμεθα, μα δεν είναι φιλοπεριβαλλοντικές στην ουσία, γιατί συνεισφέρουν ουσιαστικά, ε, συμβάλλουν στην αποψήλωση του δάσου του Αμαζονίου. Ενώ λοιπόν εμείς στη Σουηδία περηφανευόμαστε για τις φιλοπεριβαλλοντικές μας δημόσιες συγκοινωνίες κόβονται τα δέντρα του Αμαζονίου και αυτόχθονες κινδυνεύουν. Πρέπει να την αναθεωρήσουμε εκ βάθρων τη στρατηγική μας στην Ευρώπη γιατί είναι καταστροφική. Αρκεί να καταλάβουμε ότι για τα βιοκαύσιμα χρειαζόμαστε όλο και περισσότερο φινικέλαιο και αυτό θα καταστρέψει εντελώ τον Αμαζόνιο, τον πνεύμα του πλανήτη μας. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Μαρίζα Ματίας από την ΚΟΕ. Κύριε Πρόεδρε, αυτό το οποίο βλέπουμε στον Αμαζόνιο είναι μία τραγωδία. Έχουμε μία επίθεση στο περιβάλλον, στους αυτόχθονες, οι οποίοι αποδεκατίζονται και είχαν εγκαταλειφθεί στην πανδημία. Στην Βραζιλία υπάρχει ένας πρόεδρος, ο Μπολσονάρο, ο οποίος προωθεί δραστηριότητες ε, και πράξεις εγκληματικές. Μιλάμε για μια χώρα ε, της οποίας ο πρόεδρος είναι κατά του λαού του, κατά των αυτοχθόνων. Ο Επίτροπος είπε πως ε, είμαστε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει η συμφωνία με τον Μερκοσούρ. Στη συμφωνία αυτή πρέπει να ασκήσετε πίεση για να γίνουν σεβαστά αυτά τα δικαιώματα. Είμαστε ειλικρινείς συμφωνία αυτή έχει υπογραφεί τόσο καιρό δεν βλέπουμε πουθενά καθόλου καμία πίεση. Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Δεν είναι δυνατόν να ε, καταστρέφουν τον Αμαζόνιο και τους αυτόχθονες. Ε, γι' αυτό απευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ακούσει την φωνή των Βραζιλιανών, των αυτοχθόνων που υπερασπίζονται τον Αμαζόνιο. Πρέπει να είμαστε στο πλευρό των λαών και όχι των πολυεθνικών. Σας ευχαριστώ. Κυρία Σπυράκη, παρακαλώ. Οι συνάδελφοι, οι εικόνες της καταστροφής της ζούγκλας του Αμαζονίου στοιχιώνουν τη συλλογική μνήμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να έφυγαν από τις οθόνες, όμως η καταστροφή είναι εκεί. Και η κυβέρνηση της Βραζιλίας ενθαρρύνει πλέον με νόμο την αρπαγή γης που στόχο έχει την υπερκαλλιέργεια της σόγιας την υπερεκτροφή των βοηδών την υπερεκμετάλλευση του δάσους με στόχο την παραγωγή καουτσούκ. ξέρετε όλα αυτά τα προϊόντα για να παράγονται σε τόσο μεγάλες ποσότητες σημαίνει ότι διατίθενται στις αγορές και εκεί ακριβώς είναι και η δύναμή μας. Ω ευρωπαϊκή ένωση διαθέτουμε την ενιαία αγορά και οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμή μας για να δείξουμε το δρόμο είναι πολύ σημαντικό να ελέγχουμε στην πράξη τις προϋποθέσεις της εμπορικής μας σχέσης με τις χώρες της μερκοσούρ και όσο χρειαζόμαστε την εμπορική συμφωνία με τις χώρες της μερκοσούρ άλλο τόσο χρειαζόμαστε και την εφαρμογή των κανόνων της συμφωνίας του παρισιού. σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ενθαρρύνουμε πρακτικές που